Okay, colleagues, we're a little bit... Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει λίγο, διότι ήμασταν στο άλλο κτίριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο φίλος μας συνάδελφος Μωρίς Πονγκά έχει επιστρέψει και τον κάνουμε να εργαστεί πολύ σήμερα και να μετακινείται από το ένα τμήμα του κτιρίου στο άλλο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο 27 της ημερήσιας διάταξης, σύνδεση των υπερπόντων χωρών και δαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφενό και τη Γερλανδία και του Βασιλείου τη Δανία αφετέρου. Πρόκειται για μια νέα απόφαση για σύνδεση, προκειμένου να υπάρχει μια νέα απόφαση πλαίσιο για τη σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερπόντων χωρών και δαφών. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο συνάδελφο Μόχης Μπονγκά, ο οποίο είναι ειδικό στο ζήτημα αυτό, είναι και εισηγητή για το ζήτημα αυτό. Στα πλαίσια της διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 203 και τη συνθήκη, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει και τη γνώμη του Κοινοβουλίου πρωτού προχωρήσει σε απόφαση. Στη συνεδρία του Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να παρουσιάσει το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την Ένωση Πρεπόντων Χωρών και Εδαφών και ακούσαμε επίσης και την άποψη της Οκτάτης Ένωσης Ένωση Πρεπόντων Χωρών και Εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει επίση και με το σύστημα DCI, τον μηχανισμό χρηματοδότηση τη αναπτυξιακή συνεργασία, καθώ επίση σχετίζεται και με το νέο μέσο χρηματοδότηση, το ΕΝΤΙΚΙ. Δίνω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Πόγκα. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης μου όσον αφορά τη νέα απόφαση σύνδεση των υπερπόντων χωρών και δαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε το ζήτημα αυτό μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές Είμαι πραγματικά ικανοποιημένο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο ένα ειδικό μέσο το οποίο θα έχει να κάνει με, με τι περπόντιε χώρε και εδάφη. Πρόκειται για αίτημα το οποίο είχε υποβάλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι θετικό ότι θα υλοποιηθεί αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περπόντιε χώρε και εδάφη δεν είναι αναπτυσσόμενε χώρε. Είναι μέλη τη ευρωπαϊκή οικογένεια και καλούνται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερε δυσκολίε και χρειάζεται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις προκειμένου να φέρουν εις πέρας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει υπόψη στο Brexit και προβλέπει μια εταιρική σχέση για 13 πλέον υπερπόντιες χώρες και δάφη που βρίσκονται στον Ατλαντικό, την Καραϊβική, την Αρκτική, τον Ειρηνικό και τον Ειδικό ωκεανό. Η πρόταση είναι πολύ καλή ποιότητα και θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ για την πρόταση αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν και για το λόγο αυτό ακριβώ. πρότεινα 87 τροπολογίε αφού ήρθα σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών, με προσώπους των υπερπόντων χωρών και εδαφών και με, τις, με τα σχετικά κρατημέλη. Θα σας παρουσιάσω τα τέσσερα βασικότερα σημεία των προτάσεών μου. Καταρχάς, θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική διάσταση της σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και προποντίων χωρών και εδαφών. Η εταιρική αυτή σχέση είναι μοναδική και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι υπερπόντιε χώρε και εδάφη να εμπλέκονται περισσότερο στην θέσπιση ευρωπαϊκών στρατηγικών στι περιοχέ όπου βρίσκονται. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω εκπρόσωπο των Ευρωπαίων πολιτών, και ως εκπρόσωπο επομένω και των πολιτών από τι περπόντιες χώρε και δάφη θα πρέπει να συνδέεται περισσότερο με την όλη πολιτική διαδικασία. Δεύτερο σημείο. Χαίρομαι για το ότι έχουμε πλέον ένα μέσο το οποίο εντάσσεται στο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι αρκετά διαφανή η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων ανάμεσα στι διάφορε υπερπόντιε χώρε και δάφη και βλέπουμε μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό, μια χρηματοδότηση για τη Γρυλανδία, ενώ για τις 12 υπόλοιπες χώρες και εδάφη δίδεται ένα γενικό ποσό χωρίς επιμέρους λεπτομέρειες. Στην έκθεσή μου λοιπόν προτείνω η κατανομή για κάθε υπερπόντια χώρα και εδάφη να είναι συγκεκριμένη. Προτείνω συγκεκριμένα ποσοστά ανά χώρες και εδάφη, ποσοστά τα οποία είναι πιο δίκαια και βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο ενέκρινε την ανθεωρημένη προσέγγιση του όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και επομένω, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα θέλαμε να έχουμε πλέον 669 εκατομμύρια ευρώ για το μέσο αυτό και όχι 500 εκατομμύρια ευρώ, όπω προβλέπεται τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ανάγκε είναι πολύ σημαντικέ και οι υπερπόντιε χώρε και θα πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσά είναι χαμηλά και δεν μπορούμε να κατεβούμε κάτω από τα 669 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τον προγραμματισμό. Στα πλαίσια τη νέα αυτή απόφαση για τη σύνδεση θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε και δεν θα πρέπει να γίνεται συνεχώ μία παραπομπή στου κανόνε του Μηχανισμού Γειτονία, Αναπτυξιακή Συνεργασία και Διεθνού Συνεργασία. Αυτό σύγχυση μόνο προκαλεί και δεν ανταποκρίνεται στι ανάγκε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπερπόντιων χωρών και δαφών. Οι υπερπόντιες χώρες και δάφη είναι κυρίως νησιά με λίγου κατοίκους Στη Σάρτα έχουμε κάτω από 2.000 κατοίκου, στη Γουάλη και είναι 15.000. Οι κανόνε λοιπόν προγραμματισμού θα πρέπει να απλουστευθούν και να επικεντρώνονται στα πιο ουσιώδη στοιχεία. Τέλο το ζήτημα της ε, πρόσβασης στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο προτείνω ότι στα πλαίσια της απόφασης για τη σύνδεση θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταστήσει τα προγράμματα αυτά προσβάσιμα στις περπόντιες χώρες και δάφη κάνοντας, αν κρίνεται αναγκαίο, και τις απαραίτητες προσαρμογές. Για παράδειγμα, δούμε το πρόγραμμα Εράσμους. Αν δεν προσαρμοστούν να προσαρμοστεί η κάλυψη μάλλον των ταξιδιωτικών δαπανών στι ιδιαιτερότητε των υπερποντίων χωρών και δαφών που είναι πολύ πιο μακριά και επομένω η τιμή του εισιτηρίου πολύ πιο υψηλή, τότε το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει βέλτιστα για του κατοίκου αυτών των χωρών και δαφών. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίδονται οι απαραίτητε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τι υπερπόντιε χώρε και δάφη από μία αποκλειστική διαδικτυακή πύλη για τι περιοχέ αυτέ. Θα ήθελα πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων των μελλοντικών να λάβει δόντω υπόψη τι παρατηρήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι σαφέστατε αυτέ προτάσει που έκανε. Η Μαρία Ρόιγκμπουκ μα ζήτησε να πάρει πρώτη το λόγο γιατί πρέπει να πάει σε μια άλλη επιτροπή. Με τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν των υπολείπων συναδέλφων δίνω στη Μαρία πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πολυμορείς για αυτό το σχέδιο. Πρώτος, παιδιά μας πλευρά είναι ένα πολύ καλό σχέδιο όσον αφορά την Ατζέντα 2030. Ε, είναι καλύτερα τώρα το έγγραφο και ε, τα κονδύλια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την κατάσταση με την κλιματική αλλαγή. Ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει πληθυσμό που υποφέρει από ε, την αλλαγή του κλίματο. Επίση, συμφωνώ με τη διατύπωση για την ισότητα των ε, φύλων, για το gender mainstreaming, τη ένταξη τη ε, διάσταση του φύλου. Επίση όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων, ε, τη συγκεκριμένη κατανομή θεωρώ ότι αυτό θα επιφέρει διαφάνεια και είναι πολύ σημαντικό. Το μόνο που μας λείπει είναι το ερώτημα αν θα μπορέσουμε τελικά να συμπεριλάβουμε τις περπόδιες ε, ε, χώρες και εδάφη στα διαθροντικά ταμεία. Δεν αναφέρεται κάτι σχετικό μέσα στο σχέδιο της πρότασης. Θα μπορούσαμε όμως να το υιοθετήσουμε και αυτό. Και κάτι ακόμα που μας ε, προβληματίζει είναι η τροπολογία 45, γιατί θεωρούμε ότι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει στρέβλωση ε, του εμπορίου εξαιτία των ε, επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κατά τα άλλα και συγγνώμη που ε, θα πρέπει να φύγω αμέσως. Thank you, Maria. Ευχαριστώ, Μαρία. Θα ήθελαν άλλοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Uh, uh, uh, Είναι σημαντικό το θέμα. Έχουμε από τη μία πλευρά ε, τέσσερι ε, φορεί που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του οικοσυστήματο. Είναι προτεραιότητα εμπειρπόντιες χώρες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά και τη βιοπικιλότητα και τη γεωγραφική τους θέση, χρειάζονται τη στήριξη τη Ευρωπαϊκής Ένωση για να μπορέσουν να ε, προχωρήσουν σε αλλαγές όσον αφορά την μείωση τη φτώχεια. Θετικέ συνέργειες σε αυτό το πλαίσιο είναι η εστίαση που έχουμε στην οικοδόμηση ικανότητα, η αναθόρηση των διατάξεων από τότε που όλα αυτά βρίσκονται από την αιγίδα της ε, ευρωπαϊκής οικογένειας and attracting private investments from windmills, solar parks. Οπότε γίνεται λόγος πλέον για τα εργοστάσια υδροελεκτρικής ενέργειας και όπως γνωρίζετε πολλοί φορείς κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις για να πετύχουν τη μετάβαση σε μια ανάπτυξη οικονομική που θα σέβεται όμως το περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις πτυχές, έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρξει ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο και προπολογισμό που θα απευθύνεται στα OCTs. Θα απευθύνεται στι υπερπόντε χώρε και εδάφη. Η συνεργασία μεταξύ των υπερπόντιων χωρών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά που προτείνονται μέσα στι ε, τροπολογίε του κυρίου Πόγκα θεωρώ ότι είναι πολύ καλά εξορροπημένε και λαμβάνουν υπόψη και το Brexit. Οι συμφωνίε σύνδεση θα πρέπει να βασίζονται σε τρει πυλώνες, την ανταγωνιστικότητα, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την μείωση της, ε, του βάλου του χαρακτήρα. Επίσης, ε, η ένταξη και άλλων ε, εταίρων και γειτονικών περιοχών. Πρέπει αυτή η σύνδεση να βασίζεται πάνω σε ισχυρούς θεσμούς και να υπάρχει μεγαλύτερη ε, συνεισφορά στο φάκελο που αφορά την κλιματική αλλαγή. Τέλος, ήθελα να υπογραμμίσω και να τονίσω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την εστίασή μας στο να βρούμε καλύτερους τρόπους για να ε, κάνουμε την οικονομική ανάπτυξη ε, πιο επωφελή για περισσότερο αριθμό ατόμων και με στόχο να πετύχουμε τους στόχους ε, της Συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και ευχαριστώ βέβαια και τον εισηγητή μας και ελπίζω πραγματικά ότι θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε πολύ επικοδομητικά για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ήθελε κάποιο άλλο συναδέλφο το λόγο για το θέμα αυτό. Ενώ όχι, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει εκπροσωπο. Ε, δηλαδή, δεν έχω τα ονόματα σα. Κυρία Μινιό, από την Γενική Διεύθυνση Αναπτύξη και Συνεργασίας. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, είπα μέλη του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί τον κύριο Μωρή Πόγκα για το προσχέδιο έκθεση, γιατί με αυτό καλωσορίζει το προσχέδιο απόφαση της Επιτροπή και αναφέρει και σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η σχέση μας με τις υπερπόντιες χώρες και περιοχές. Θα σταθώ τώρα σε ορισμένα από τα στοιχεία που, ζητήματα που θέτει η έκθεση. Το πρώτο είναι το θέμα της μεγαλύτερης συνεργασίας ε, στο πολιτικό επίπεδο. Η Επιτροπή συνεχίζει να επιθυμεί τον πολιτικό διάλογο με τις υπερπόντιες περιοχές. Αυτό το νομικό πλαίσιο θα μας δώσει την δυνατότητα να λαμβάνουμε δράση και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώκει να έχουμε μεγαλύτερο πολιτικό πιο και πιο συχνό πολιτικό διάλογο με αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα για το ζήτημα της περιφερειακής τους ανάπτυξης και εξάλλου στις αρχές του 2019 θα οργανώσουμε και ένα φόρουμ για να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους όλων αυτών των περιεχών. Θα υπάρχει εκπροσώπηση βεβαίω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Προεδρίας του Συμβουλίου σε αυτό το ετήσιο φόρουμ. Δεύτερον, λέγεται ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί το εργαλείο αυτό στις ιδιαιτερότητες κάθε ε, υπερπόντιας χώρας. Καταγράφουμε τις ανησυχίες που εκθέτει ο εισηγητής σας, γιατί υπάρχουν διαφορές και θα πρέπει να σεβαστούμε και τις διατάξεις του NCDI. Ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να απλοποιήσει το το, τα εργαλεία που έχουμε και να έχουμε ένα ενιαίο προγραμματισμό που είναι αυτός που δημιουργείται με το, το εργαλείο ενδίκη. Πράγματι, ίσως να μην είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό όπως το αναφέρετε βλέποντας μόνο το εργαλείο για τις υπερπόντιες περιοχές, αλλά αυτό είναι απαραίτητο για την, για την ασφάλεια δικαίου στο μέλλον σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι έχουμε το ενδίκη θα μας επιτρέψει να ακολουθήσουμε μια απλοποιημένη διαδικασία για τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων μας σε συνεργασία με τις περπόντιες περιοχές. Μετά, το τρίτο σημείο που θέλετε, ε, η κατανομή των κονδυλίων. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τον εισηγητή εδώ. Βέβαια, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Και θα χρειαστεί να βρεθούν διάφορε συμβαστικέ λύσει. Θεωρούμε ότι δεδομένου του Brexit, τα 500 εκατομμύρια για αυτέ τι 12 υπερπόντιε περιοχέ είναι ένα εύλογο συμβιβασμό. Ε, ο ορισμός της περπόντιας περιοχής ή περιφέρειας ε, αναφέρεται στην ιστορική σχέση που μπορεί να έχουν αυτές οι περιοχές με κάποια χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου θα γίνει και μια αξιολόγηση εκ των υστέρων ε, επί τη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, των διαφόρων ε, προγραμμάτων δηλαδή, ο εισηγητής προτείνει στα κριτήρια να προτείνουμε, να προσθέσουμε μάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μας φαίνεται ορθό δεδομένου ότι όλες οι υπερπόντιες περιοχές πλήττονται από την κλιματική αλλαγή. Μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως βασική της αρχή ότι οι προτάσεις θα είναι καταρχήν επιλέξιμες όταν προέρχονται από αυτές τις περιοχές. Το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση έρχεται από υπερπόντια περιοχή ή χώρα για οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο θεωρείται καταρχήν επιλέξιμη, καταρχήν δεκτή σαν να προερχόταν από κράτους μέλος δηλαδή. Θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για, για λόγους ασφάλειας δικαίου, έτσι ώστε να έχουμε και πιο μεγαλύτερη συμμετοχή. Τα προγράμματα αυτά θα, θα με μεγαλύτερη ε, ακρίβεια ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία οι υπερπόντιες περιοχές θα μπορούσαν να υποφεληθούν ε, από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα. Έχουμε επίσης και την ε, Ένωση των υπερπόντιων Περιοχών που θα εξετάσει και θα ενημερωθεί καλύτερα για τα διάφορα επιπλέον κριτήρια. Τώρα, αναφερθήκατε επίσης στη σημασία που έχουν οι στόχοι μας, δηλαδή η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, βιώσιμη ανάπτυξη και ε, ισότητα των φύλων. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, μια προκαταρκτική αξιολόγηση μας δείχνει ότι στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης το 23% των κονδυλίων 2014-2020, το οποίο, βέβαια, για, το, οποίο βέβαια ο προγραμματισμό δεν έχει ακόμα κλείσει, το 23% αυτών των χρημάτων πηγαίνει για δράσει για την κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τι πόντιε περιοχέ για να επιτύχουμε τους στόχους που έχει θέσει για την κλιματική αλλαγή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό θα είναι δύσκολο εάν συνεχίσουν ορισμένες από αυτές τις περιοχές να επιλέγουν τη χρηματοδότηση αυτή να κατευθύνουν προς έναν συγκεκριμένο τομέα και όχι να βλέπουν συνολικά την καταπολέμηση και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουν για την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πονγκά. Σας απευθύνθηκαν κάποιες ερωτήσεις από τη Μαρία Χόρμπερκ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν μπορείτε να απαντήσετε. Θα απαντήσω κυρία Πρόεδρε λέγοντας ότι οι υπερπόντιες χώρες και δάφοι δεν μπορούν να επωφελθούν από τα δευτικά προγράμματα που απευθύνονται στις ευρωπαϊκές περιοχές εξαιτίας του καθεστώτο τους. Είμαστε συνδεδεμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα ειδικό καθεστώ που δεν μα επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στα διαρθρωτικά προγράμματα. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι διαφορετικά για τα DOM-TOM, γιατί αυτές οι περιοχές, οι DOM-TOM, θεωρούνται ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές που ανήκουν όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι πρεπόντιες χώρες και εδάφη, τα OCTs, είναι περιοχές που είναι απλώς συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Θα διαβιβάσουμε τι απαντήσει σα στη Μαρία που χρειάστηκε να φύγει. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 22 Νοεμβρίου, ήδη λοιπόν την 5η. Πιέζει ο χρόνο όπω καταλαβαίνετε. Γιατί πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε όλε αυτέ τι προτάσει που άπτονται του πολιετού δημοσιονομικού πλησίου. Δεν λέει εδώ πέρα ποια ώρα. Μέχρι τι 12 το μεσημέρι. Ούτε καν στι 5 το απόγευμα. 5, 5 το απόγευμα. Πολύ ωραία. Ορίστε, σα δίνουμε μερικέ ώρε παραπάνω. 5 το απόγευμα, 22 Νοεμβρίου, είναι η καταληκτική προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Και θα πρέπει βέβαια να ψηφίσουμε το Δεκέμβριο, γιατί αν το κάνουμε αυτό, δεν θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε καθόλου τι συζητήσει που γίνονται στο Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε και τον κύριο Πόγκα. Α περάσουμε τώρα στο σημείο 28 τη ε, ημερήσια διάταξη εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Έχουμε την συμβολή μας τώρα στην έκθεση από την Επιτροπή Εμπορίου για την ενδιάμεση αναθεώρηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Και όπως ξέρετε το σύστημα αυτό επιτρέπει στις πιο ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες να πληρώνουν χαμηλότερους δασμούς ή καθόλου δασμούς κατά τις εξαγωγές τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι έχουν πρόσβαση προνομιακή στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί τι επιπτώσει του συστήματο αυτού, προσπαθώντα να δει πώ επωφελούνται τελικά κυρίω οι χώρε που συμμετέχουν στο λεγόμενο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων PLUS, χώρε δηλαδή που επωφελούνται ακόμα περισσότερο όταν εφαρμόσουν συγκεκριμένε συμβάσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα, συμβάσει των Ηνωμένων Εθνών, συμβάσει του, Διεθνού Οργανισμού Εργασία και έχουν πιο προνομιακή μεταχείριση οι χώρες αυτές εφόσον επίσης ε, εφαρμόζουν ε, προγράμματα που ατηρούν το, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ο κύριος Έγγελ θα πάρει το λόγο αντικαθιστώντας κανονικά τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως ε, θα γίνει δήμαρχος του Κίλ στην Πολωνία σε δύο μέρες ο μα. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω για την όλη εργασία που έκανε εν γέννη και ιδίω για τον φάκελο αυτόν. Ο κύριος Μπόγκταν Μπρούνον Βεντά έχει ήδη καταθέσει ένα κείμενο. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να κάνω αυτή τη στιγμή είναι επισημάνω δύο-τρία σημεία τόσο το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων όσο και το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων πλάσα και ιδίω το καθεστώς όλα εκτός από όπλα έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις. Όντως οι χώρες αυτές καταφέρουν και εξάγουν περισσότερο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνεται κατά αυτόν τον τρόπο η οικονομική τους ανάπτυξη και συμβάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο στην εξάλληψη της φτώχειας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το 2016 περίπου 63 δισεκατομμύρια ευρώ, μάλλον εμπορεύματα αξία 63 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των προτιμήσεων του σίγμα γάμα πι εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε όμως ότι δεν λειτουργούν όλα τα μέσα με τον ίδιο τρόπο ούτε έχουν τις ίδιες επιπτώσεις. Έχουμε 31,6 δισεκατομμύρια ευρώ από δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων και έχουμε μόνο 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ από δικαιούχους του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων Plus και 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ από δικαιούχου του προγράμματο Όλα εκτός από τα όπλα, που σα κάνει και οι πιο φτωχέ χώρε του πλανήτη. Για το SPG+, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. Το επίπεδο αιρεσιμότητας πολύ υψηλό, επομένως 8 μόνο είναι χώρες οι οποίες είναι επιλέξιμες και μία μόνο χώρα βρίσκεται στην Αφρική. Νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε στο μέλλον να δούμε πώς θα μπορούσαμε να διευρύνουμε κάπως το πρόγραμμα αυτό και προς άλλες χώρες οι οποίες από οικονομικής πλευράς βρίσκονται στο ίδιο πάνω κάτω επίπεδο αλλά οι οποίες δεν είχαν καταφέρει μέχρι στιγμής να τηρήσουν όλα τα κριτήρια ρεσιμότητος τα οποία έχουμε επιβάλει εμείς. Λέγοντας βέβαια ότι έχει γίνει σαφής πρόοδο από τις χώρες που συμμετέχουν στο SPG+, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος καθεξής. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο όντας γνωμοδότηση είναι και ένα κείμενο αρκετά σύντομο και εν γέννη βέβαια η αποτίμηση είναι αρκετά θετική. Ελπίζουμε να μην υποβαθμιστεί η σημασία αυτού του μήνυματος που είναι πολύ ξεκάθαρο. Έχουμε τους κοιόδες εισηγητές. Ο Ντόναβαν, λόγω σε σένα. Είναι τιμή μου να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί σας εδώ στην πιο, μια από τις πιο σημαντικές επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Το ε, σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων δημιούργησε ε, ένα σύστημα δασμών λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, την ε, καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Μια διάμεση αξιολόγηση που έγινε Μπορώ να πω ότι η Επιτροπή με αυτή την έκθεση έκανε μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την λειτουργία και τα αποτελέσματα του συστήματος γενικευμένων προτεμήσεων. Είναι θετική η επιρροή στην αύξηση των εισαγωγών που αποτελούν το 5% των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια οριακή αύξηση στην εξαγωγή των 23 χώρων που συμμετέχουν στο σύστημα αυτό από το 2014. Η αύξηση στην χρήση ε, τη φορολογική αυτή διευκόλυνση αφορά εξαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων είναι ένα βασικό εργαλείο κλειδί για την ανάπτυξη και πρέπει να συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο. Γι' αυτό η ενδιάμεση αυτή έκθεση μας παρέχει ευκαιρίες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το μηχανισμό αυτό στο μέλλον. Για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια η έκθεση δείχνει ότι αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Η Επιτροπή πρέπει να δείξει προθυμία να αναλάβει δράση όταν οι χώρες μένουν πίσω στις δεσμεύσεις τους ή όταν δεν ε, σημειώνεται σημαντική πρόοδος. Βλέπουμε θετικά ε, την δράση για έρευνες που έγινε στην Μιανμάρ και στην Καμπότζη και αυτό είναι κάτι πρέπει να το τονίσουμε γιατί είναι μεγάλη σημασία του εφόσον βλέπουμε χώρες όπως το Βιετνάμ να συνάπτουν ε, ε, συμφωνίες ελευθερία μπορεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμφωνίες ελευθερία μπορεί είναι πολύ πιο δύσκολο να αναστολούν εξαιτία ε, παραβίαση των δεσμεύσεων. Γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία ε, υπό το πλαίσιο, στο πλαίσιο των, γενικευμένων προτιμήσεων. Είναι κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε και να εφαρμόσουμε ε, τη σύμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Δεν μπορεί το σύστημα αυτό να επιλέξει όλα τα προβλήματα, αλλά σίγουρα είναι ένα εργαλείο πολύ αποτελεσματικό ε, για την μείωση της φτώχειας. Η απελευθέρωση του εμπορίου από μόνη της δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Το σύστημα έχει αυξήσει το εμπόριο για τις χώρες εταίρους και υποστηρίζει την δίκαιη κατανομή του πλούτου που προκύπτει από αυτό υποστηρίζει την ε, διαφοροποίηση και την ισότητα και αποτρέπει την ε, αρπαγή γεών. Επίσης, διευκολύνει και την κοινωνική ανάπτυξη και την διασφάλιση των ανθρωπίνων ε, γερασιακών δικαιωμάτων και ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία πάνω σε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Um, thank you very much. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο στο σημείο αυτό της μέσης διάταξης. Αν όχι, ε, θα θέλαμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, ο κύριος Χάτουμ, την DigiTrade. Δεν ξέρω αν το έχω προφέρει στο όνομά σα. Thank you, Chair. Yeah, that's enough. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Σας ευχαριστώ που προσπαθήσατε να προφέρετε στο όνομα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση. Πιστεύω ότι είναι ε, θετική η έκθεση. Εξάλλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ε, σύνταξη, στο να συντάξουμε αυτόν τον κανονισμό. Μία από τα, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της αξιολόγησης είναι ότι το σύστημα δουλεύει εάν συγκρίνουμε τι συνέβαινε πριν και τι συνέβαινε μετά. Και αυτός ήταν ο στόχος του κανονισμού. Έχουμε στοιχεία. Το πρόγραμμα όλα εκτό από όπλα είναι το πιο γενναιοδέρο και εδώ έχουμε ένα 62% αύξηση των εξαγωγών και στο GSP Plus αύξηση 54%. Σημαντικό είναι επίσης να επισημάνουμε ότι αυτά τα προγράμματα δεν πλήττουν τη δική μας βιομηχανία. Ακριβώς επειδή φροντίσαμε να θέσουμε κριτήρια και η εισαγωγές μπορεί να μειώνονται αλλά κατανέμονται σε εκείνες τις χώρες που τα χρειάζονται περισσότερο αυτά τα εμπορεύματα. Υπάρχουν ζητήματα σε ορισμένες από αυτές τις χώρες που έχουν σχέση με την διακυβέρνηση, με τους θεσμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να πει κανείς τι πρέπει να γίνει είναι ίσως ανεκδοτολογική, περιπτωσιολογική η περιγραφή που δίνεται σε, σε για ορισμένες χώρες. Ίσως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε επ' αυτού για να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού και διαπιστώνουμε ότι η συμμετοχή των κρατών μελών θα μπορούσε να βελτιωθεί, να ενισχυθεί. Θέλουμε να το προωθήσουμε αυτό από την πλευρά της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής. Ήδη προσπαθούμε να εμπλέξουμε περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κανονισμός για να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι ακόμα πιο σημαντικό να υπάρξει αξιοποίηση αυτού του συστήματος στις χώρες δικαιούχους. Ε, παρά το γεγονό ότι έχει αυξηθεί η χρήση του συστήματος, είναι σημαντικό να δούμε αν μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης και έναν μηχανισμό για να αποχωρεί μια χώρα από το σύστημα GSP, ε, τίθεται ένα ζήτημα αξιοπιστία. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιείται και αυτός ο μηχανισμός όταν πρέπει για λόγους αξιοπιστία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί μάλιστα να έχουμε και ε, ουσιαστική παρέμβαση και ουσιαστικές αλλαγές να πετύχουμε σε ορισμένες από αυτές τις χώρες η σχέση ανάμεσα στην αναπτυξιακή συνεργασία και το GSP είναι προφανής, αλλά νομίζω θα έχει νόημα να την δούμε περισσότερο στην πράξη. Εξάλλου, ένας από τους στόχους του GSP ή του GSP Plus είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εξαγωγών των χωρών δικαιούχων. Δηλαδή να υπάρξουν επενδύσει, να υπάρξει μια διευκόλυνση τη οικονομία του, ε, έτσι ώστε να αρχίσουν να εξάγουν και σε περισσότερου τομεί από ό,τι στο παρελθόν. Ε, στην έκθεση βλέπουμε ότι έχει συμβεί αυτό, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Είναι λοιπόν ένας τομέας εδώ που θα μπορούσαμε να τον δούμε περισσότερο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί κανόνες για την προέλευση των προϊόντων, στους οποίους θα πρέπει να τηρεί κανείς για να αξιοποιήσει το προτιμησιακό καθεστώς και αυτό ίσως δυσκολεύει ιδιαίτερα τις μικρότερες και φτωχότερε χώρες η τήρηση των τελωνιακών κανόνων. Τέλος, γνωρίζετε ότι η πολιτική μας οφείλει να βασίζεται σε αρχές. Πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι καινούρια φιλοσοφία, ε, ε, διαφορετική φιλοσοφία από αυτό με το οποίο έχουν συνηθίσει ορισμένες από αυτές τις χώρες εταίροι ε, δηλαδή το ότι συνδέουμε το διεθνές εμπόριο με κάποιες άλλες αξίες. Και νομίζω ότι αυτό ε, προσπαθούμε να τους το εξηγήσουμε και, ότι, ε, και πιστεύουμε ότι βεβαίω είναι εφικτό να δημιουργήσει κανεί μια διεθνή οικονομία και ένα διεθνέ εμπόριο το οποίο παράλληλα να βασίζεται σε αρχέ. Θέλουμε να υπάρχει Πλήρη εμπλοκή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Κοινωνία των Πολιτών ε, και των κρατών μελών έτσι ώστε να βελτιώσουμε την εφαρμογή αυτού του συστήματο και ακριβώ αυτό θα πράξουμε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζοντα τα ευρήματα τη εκθέση αυτή. Σα ευχαριστούμε πολύ λέει και η πρόεδρο. Πράγματι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς η Επιτροπή του Κοινοβουλίου μπορεί να εξετάσει το ζήτημα αυτό, δηλαδή πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις χώρες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνονται μέσω του προτιμουσιακού καθεστώτος και ίσως με μια τροπολογία να το αναδείξουμε περισσότερο. Ο Φραγκέγγελς, δεν νομίζω ότι επί της ουσίας μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξίας, θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης και εν τέλει αυτός είναι από τους τομείς όπου εμείς μπορεί να πετύχουμε τελικά τους στόχους μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προσπαθώντας να αυξήσουμε πολύ έντονα ένα εμπόριο το οποίο να είναι οικονομικά υποφελές για τις χώρες που συμμετέχουν στην πολιτική ε, αναπτυξιακή συνεργασία στην οποία προωθούμε. Θα πρέπει δηλαδή να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διευρύνουμε την χρήση και το πεδίο εφαρμογής όλων αυτών των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου τα μέσα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερες τρίτες χώρες. Πολύ ωραία, σα ευχαριστούμε πολύ. Προβλέπετε μια, μια άλλη προθεσμία αυτή τη στιγμή για την κατάθεση τροπολογιών 30 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί. Έχετε περισσότερο χρόνο. Θα ψηφίσουμε 21-22 Ιανουαρίου. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη συνεδρία στο ζήτημα αυτό με την παρουσία εκπροσώπων από την Επιτροπή Πολιτισμού. Έχουμε μαζί μας πάλι την συντάκτρια γνωμοδότηση, την Ελένη Θεοχάρους, η οποία αυτή την εβδομάδα έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά για την Επιτροπή μας. Θα ήθελα λοιπόν να σε υπενθυμίσω ότι ε, μέρος της ε, πρότασης αυτής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να καταφέρουμε να έχουμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αλλά να καταφέρουμε επίσης να το συνδυάσουμε και με την πρωτοβουλία θελοντική ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεφάλαιο 4 είναι δική μα αποκλειστική αρμοδιότητα, ενώ τα κεφάλαια 6, 7 και 8 είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπή Πολιτισμού. Άρα δεν μπορούμε εμεί να έχουμε τροπολογίε για τα κεφάλαια αυτά. Τα άρθρα μάλλον 6, 7 και 8 δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τροπολογιών για τη δική μα την Επιτροπή ή αν έχετε τι τροπολογίε πρέπει να τι προωθήσετε κατευθείαν στην Επιτροπή Πολιτισμού. Για όλα τα υπόλοιπα άρθρα έχουμε συντρέχου αρμοδιότητα. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην συντάκτρια γνωμοδότηση Ελένη Θεοχάρου για να μα παρουσιάσει την γνωμοδότηση αυτή. Έχετε το λόγο, Ελένη. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρωτού παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να πω ότι το σκληρό, σκληρή δουλειά έγινε από την συνάδελφό μου, τη Χαριτίνη Μιχαηλίδου και είναι σωστό να το αναφέρω. Εξ αρχής ήμουν της άποψης ότι εξέφρασα τις απόψεις μου στο διάλογο που είχαμε τις προάλλες. Θεωρώ η συγχώνευση της ε, πρωτοβουλίας ε, ανθρωπιστικής βοήθειας με το σώμα αλληλεγγύης μπορεί να είναι κάτι πολύ θετικό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και ενδεχομένω είναι η λύση. Και αν το προωθήσουμε σωστά θα αποτελέσει εφαλτήριο για αυτούς που ενδιαφέρονται για τον ανθρωπιστικό τομέα και σημείο εισόδου στον εθελοντισμό. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατόν για ε, μη κερδοσκοπικέ ε, οργανώσεις να, και άτομα να αποφοληθούν από δυνατότητες εκπαίδευσης ε, με τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα. Γι' αυτό το λόγο η σύστασή μας δεν είναι να εφαρμόσουμε τον το όριο ηλικία των 30 ετών. Είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα ε, στο πλαίσιο των θελοντών αλλά να δεχόμαστε και πιο πεπειραμένα άτομα να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους η πρότασή μας ζητάει να διατηρηθεί το όριο ηλικία για το σώμα, όμως η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων πάνω από αυτό το ηλικιακό όριο θα μπορεί να δικαιολογηθεί για το σώμα αλληλεγγύης. Επίσης θα είναι δυνατόν για επαγγελματίες και οργανώσεις να επιφελθούν από προγράμματα εκπαίδευση σε περίπτωση που θα θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά. Είναι σημαντικό ότι οι οργανισμοί που έχουν ήδη εμπιστευτεί δεν θα πρέπει να περάσουν την ίδια διαδικασία εκ νέου εφόσον θα τεθεί σε ισχύ ο νέο κανονισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν δηλωθεί. Επιπλέον, οι απλουστευμένε και βελτιστοποιημένε διαδικασίε και το νέο σήμα ποιότητα είναι πολύ σημαντικά για του συμμετέχοντε οργανισμού. Ακόμα η Επιτροπή μα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διατάξει ε, που αφορούν το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστική Βοήθεια είναι σύμφωνε και συμπληρωματικέ ω προ τι άλλε δραστηριότητε ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και με την ανθρωπιστική βοήθεια όπω ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Αντίληψη. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις ανθρωπιστικές αρχές και να υπάρξει συντονισμένη και αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι τροπολογίες που προτείνονται εστιάζουν στην ε, ανάπτυξη οργανικών και τοπικών ικανοτήτων, στην ανεφικτικότητα, ε, στην αποκατάσταση που θα αντιμετωπίζουν τη σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστική βοήθεια και ανάπτυξη. Εστιάζουν επίση στη μείωση του κινδύνου καταστροφών και γενικότερα την ευαισθητοποίηση και την επικοινωνία σχετικά με τι ανθρωπιστικέ ανάγκε και αρχέ. Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη στην αρχή, να μην αφήνουμε κανέναν πίσω, να του φροντίζουμε όλου, να εστίασε επίσης την εξάλληψη τη φτώχεια στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φίλων. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην πρότασή μας. Ένα τελευταίο σημείο. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές διατάξεις του προτινόμενου κανονισμού, η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα ε, ποσά για κάθε ε, κλάδο. Ο συνολικός φάκελος στην εφαρμογή του προγράμματος, στο σύνολό του, θα είναι 1 δισεκατομμύριο 260 εκατομμύρια ευρώ με τις τρέχουσες τιμές. Θα πρέπει να το αναλογιστούμε αυτό περισσότερο για να έχουμε μία πρόταση η οποία αποτελεσματικά θα αντιμετωπίσει την κατανομή των κονδυλίων για το σώμα αλληλεγγύης. Θα, θα προτείνω τροπολογίε για το θέμα αυτό και επίσης ε, ευπρόσδεκτες είναι και οι προτάσει από του συναδέλφους μου και από τους σκιώδει συζητητές. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Some of the... Και εμεί σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γερέρο είναι, όχι, ο κύριος Σένφιλτ είναι παρόν, είναι ο Άνταμε και αυτός παρόν, σκιώδης από το ΕΛΚ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Mogę właściwie mm, same dobre słowa. Λοιπόν, ε, μόνο καλά λόγια έχω να πω για το φάκελο αυτό. Και είμαι ιδιαίτερο ευτυχή γι' αυτό. Η εισηγήτριά μα έχει καλύψει το θέμα εξαντλητικά, το ίδιο και όλοι οι συνάδελφοι και νομίζω ότι η έκθεση που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ καλού επίπεδου. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν και πολλές τροπολογίες, είναι τόσο καλό το κείμενο δηλαδή, ήδη. Και ε, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο στην ε, προσπάθεια αυτή είναι οι στόχοι που θέτουμε. Το πρώτο ζήτημα, το ανέφερε και η κυρία Θεοχάρους, είναι το όριο ηλικίας συμφωνώ μαζί της, δεν χρειάζεται. Ε, δηλαδή το όριο ηλικία δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι οι στόχοι που θέλουμε να επιτυγχάνει, να αυτό το σώμα. Επομένως, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σώμα ευρωπαϊκό, ισχυρό, επαγγελματικό, εάν θέλουμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο στην Ευρώπη για να παρεμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, ε, και αν θέλουμε οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται εθελοντικά μεν αλλά με υψηλό επίπεδο δε, τότε πιστεύω ότι δεν χρειάζεται, θα ήταν λάθος μάλλον, να θέσουμε ένα όριο ηλικίας. Δεν έχει νόημα να βάλει κανείς ένα τέτοιο όριο ηλικίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι αποτελεσματική η παρέμβασή μας, το έργο αυτής, αυτού του σώματος. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η ε, ηλικία των εθελοντών που θα το ε, επιτελούν. Το ζήτημα είναι να γνωρίζουν το αντικείμενό τους, να μπορούν να κάνουν καλά ε, τη, τη δουλειά τους. Ε, εξάλλου, όπως είπατε κι εσείς, θα μπορέσει να λειτουργήσει και σε μια μορφή μαθητείας για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό, μέσω αυτού του σώματος να μάθει και να γνωρίσει το τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στα περισσότερα κράτη-μέλη ορίζουμε τον νέο ως έναν άνθρωπο κάτω των 35 ετών. Αν δείτε όμως την πραγματική ηλικιακή κατανομή των εθελοντών, ε, έχουμε από όλες τις ε, ηλικίες, από 18 μέχρι 50. Γι' αυτό συμφωνώ και με την εισηγήτρια ότι το, ε, όριο ηλικίας θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Αφού αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η αποτελεσματικότητα. Και αυτό είναι το δεύτερο το οποίο θέλω να σημάνω, είναι ότι τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο, όχι για αν θέλετε, σκοπούς δημοσιότητας, δεδομένου μάλιστα ότι ότι ε, δεν έχουμε και πάρα πολλά χρήματα στη διάθεσή μας. Λέμε ότι θέλουμε να φτάσουμε τους 100.000 εθελοντές μέχρι το 2020. Ε, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο να το πετύχουμε αυτό εάν δούμε τον τρόπο με τον οποίο προωθούμε το σώμα αυτό σήμερα. Εξάλλου χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να, για τους οποίους να μπορούμε να ανακοινθούμε την ασφάλεια τους. Δεν θέλουμε να βρεθούμε με κάποιους ίσως πολύ νέους εθελοντές που δεν γνωρίζουν ακριβώς που πηγαίνουν και μπορεί να βρεθούν και σε επικίνδυνες καταστάσεις. Ε, ε, Επομένω, προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω θα πρέπει να αναλάβουμε περισσότερη δράση, να σκεφτούμε εάν εδώ χρειάζεται κάποια τροπολογία για να το αναδείξουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Μετά, πρέπει να αναφερθούμε στη σημασία που έχει η συνεργασία με χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που αυτή τη στιγμή αναλαμβάνουν παρόμοια προγράμματα. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία. Κατά τα άλλα, για τον προϋπολογισμό, για τη δομή του προϋπολογισμού έχουμε τη βασική δομή. Για τις λεπτομέρειε του προπολογισμού, νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν είναι ανάγκη να το συζητήσουμε σήμερα. Αυτέ είναι οι παρατηρήσει κατά την άποψή μου. Όπω σα είπα, δεν θα χρειαστούν και πολλέ τροπολογίε, γιατί η έκθεση είναι ήδη πολύ καλή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριο Γερέρο. Συμφωνώ με την αξιολόγηση που έκανε ο κύριος Σιένφελτ για την πρόταση αυτή. Η Ελένη νομίζω έχει περιγράψει την συζήτηση με ακρίβεια σε προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε και σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι η πολιτική μου ομάδα βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνη που περιγράφει στην έκθεσή της η Ελένη. Μιλούμε για αυτή την συγχώνευση των εθολοντών και της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως τονίζοντας ότι όταν έχουμε εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να τηρούν τις βασικές αρχές ουδετερότητα, μη παρέμβαση, ε, ανεξαρτησία, τις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας δηλαδή. Και βλέπω επίση με χαρά ότι ορισμένα από τα στοιχεία που είχα αναφέρει σε προηγούμενη ε, μας ε, συνάντηση έχουν καταγραφεί. δεν γνωρίζω εάν έχει και τόσο πολύ νόημα να θέσουμε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, να αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, μιας και εδώ πρόκειται για μια γνωμοδότηση, ενώ συνήθως τα θέματα του προϋπολογισμού ακολουθούν άλλες διαδικασίες, από άλλες επιτροπές, από την ε, Ολομέλεια, με τις διαπραγματεύσεις κτλ. Μην Κάνουμε απλώς ένα ευχολόγιο εδώ, μην, μην αναφερθούμε λίγο με wishful thinking σε έναν αριθμό εδώ. Χρειάζεται βέβαια να το αναφέρουμε σε μια παράγραφο, ξεκάθαρα, ότι χρειάζεται η απαραίτητη πόρη για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους που θέτουμε και ότι για να συμβεί αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Θέλοντων θα πρέπει να έχει περισσότερους πόρους, να αποκτήσει περισσότερους πόρους στη διάθεσή του, ε, περισσότερους από αυτούς που μέχρι σήμερα είχε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα θα χρειαστεί περισσότερους πόρους. Τώρα για το ζήτημα της ηλικία, που είναι ένα θέμα που έρχεται και ξανάρχεται. Ε, είμαι λίγο αμφίθυμος. Γιατί, απ' τη μια προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τους νέους. Να κάνουμε τους νέους να ασχοληθούν περισσότερο με ευρωπαϊκές αξίες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η συνεργασία και το να προσφέρεις βοήθεια σε μια ανθρωπιστική καταστροφή, σε μια φυσική καταστροφή. Και υπ' αυτή την έννοια έχει αξία να προσπαθήσουμε να πρημοδοτήσουμε τη συμμετοχή νέων εθελοντών, νέων, νέων, ηλικία εθελοντών. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε ότι κάποιες από αυτές τις δραστηριότητε που πρέπει κανείς να αναλαμβάνει αμέσως μετά από μια κρίση χρειάζεται, χρειάζονται εμπειρία, χρειάζονται γνώση και επίσης χρειάζονται και μια οριμότητα προσωπική ε, που δυστυχώς δεν τη βρίσκουμε εύκολα σε πολύ νεαρής ηλικίας ανθρώπους. Για αυτόν τον λόγο εγώ θα έλεγα να βρούμε μια μέση λύση. Δηλαδή, να αυξήσουμε το όριο ηλικίας, συμφωνώ, και εγώ ότι αυτό το όριο των 30 ετών είναι υπερβολικά χαμηλό. Ε, δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, να το πάμε πολύ ψηλά, αλλά το 35 μου φαίνεται λογικό. 30 είναι υπερβολικά χαμηλό, 35 μου φαίνεται λογικό επισημένοντας όμως ότι για συγκεκριμένες περιπτώσεις, για συγκεκριμένες δράσεις που μπορεί να χρειάζονται ιδιαίτερη γνώση ή εμπειρία, θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσει για να μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε και αυτούς και τη γνώση τους και την εμπειρία τους. Έτσι νομίζω ότι θα γίνει πιο σαφής η πρόταση. Ε, θα υποβάλω μάλλον μια σχετική τροπολογία. Η πολιτική μας ομάδα επίσης ε, υποστηρίζει την προσπάθεια που γίνεται να αναφερθούμε στην, ε, στην ισότητα των δύο φύλων, στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τις ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρία, και άλλες δηλαδή ομάδες, όχι μόνο το ζήτημα, να διδείξουμε το ζήτημα του φίλου αλλά και άλλες ομάδες. Γιατί θέλουμε να πούμε ότι και να γνωρίσουμε μάλλον ότι πολύ συχνά στην ανθρωπιστική βοήθεια διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά σε σε αυτήν και το βλέπουμε ακόμα περισσότερο όταν φεύγουμε από τις αναπτυγμένες χώρες και πηγαίνουμε σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Τώρα, στην γνωμοδότηση νομίζω θα μπορούσαμε να επισημάνουμε, να προτείνουμε μάλλον, να γίνει μια καταγραφή, μια απογραφή εθελοντών που έχουν ήδη συμμετάσχει σε αποστολές ή δράσεις και έτσι να δημιουργηθεί ένας κατάλογος ανθρώπων στους οποίους θα μπορούσε κανείς να απευθυνθεί και να τους καλέσει να, για να αξιοποιήσει την εμπειρία που μπορεί να αποκόμισαν από προηγούμενες τους ε, δραστηριότητες τέτοιες. Δεν είναι ο στόχος να, κάνουμε, να επαγγελματικοποιήσουμε τον εθελοντισμό και τη βοήθεια. Αλλά αν γνωρίζουμε ότι κάποιος έχει ήδη συμμετάσχει σε μια τέτοια δράση, γνωρίζει κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει υπάλληλο της ε, ανθρωπιστικής έτσι, δράσης, αλλά χρήσιμο είναι να έχει κανείς έναν κατάλογο με τους ανθρώπους που έχουν ε, συσσωρεύσει εμπειρία στο πεδίο. και να μπορέσει να συνεννοηθεί και να συνεργαστεί και με άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσει στο πεδίο σας. Ευχαριστώ. Δεν θέλουν άλλοι συναδέλφοι να πάρουν το λόγο. Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα στην Επιτροπή. Πρώτο απαντήσουν ε, το θέμα της ηλικία. Όταν συνδυάζουμε δύο διαφορετικά προγράμματα και οι συναδέλφοι το σχολείο, σαν όταν αφορά νέους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν εθελοντικά στην ανθρωπιστική βοήθεια. Συγκεκριμένα όμω υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερε ηλικίε που στο τέλο τη καριέρα του θέλουν να προσφέρουν εθελοντικό έργο και είναι ένα διαφορετικό είδο εργασία. Είμαι λοιπόν. Ε, γνωρίζω ότι βλέπουμε ότι στέλνουμε πολλά άτομα σε χώρες για να επιτελέσουν ένα έργο που θα μπορούσαν ντόπιοι νέοι σε ηλικία να αναλάβουν. αν είναι 18, 19, 20, ίσως θα μπορούσαμε πιο πολύ να το συμπεριλάβουμε σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής ή στην εκπόνηση κοινών προγραμμάτων. Γιατί να στείλουμε από εδώ νέους σε μια φτωχή χώρα, σε ένα φτωχό χωριό στην Αφρική να φτιάξουν π.χ. ένα σχολείο ενώ μπορούν εντόπιοι που μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι κάτι πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Έχουμε δει διαφορετικά πράγματα σε ένα πρόγραμμα. Πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το μήνυμα που θα θέλουμε να δώσουμε. Γιατί στέλνουμε Ευρωπαίους πολίτες στις χώρες αυτές αντί για ντόπιου που θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά. Είναι κάπως περίεργο αυτό. Επίσης, κατά πόσο στηρίζουμε οικονομικά αυτούς τους εθελοντές Σήμερα είναι η Παγκόσμια ε, Μέρα Παιδιών για τη, UNICEF. Δεν υπάρχουν προγράμματα που να δίνουν προνόμια σε άτομα που ήδη έχουν όμως και τα χρήματα και τις συνδέσεις. Είμαι κάπως... δεν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, ποιοι είναι οι νέοι που μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, πώς μπορούμε να τους βρούμε είναι συγκεκριμένα σχόλια από τα οποία αποφυτούν, υπάρχουν κάποια δεδομένα κοινωνικο-οικονομικά. Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν, που συμμετέχουν θελοντικά στα υπάρχοντα προγράμματα. Δεν θα ήθελα να καταλήγουν εκεί μόνο άτομα τα οποία έχουν τις διασυνδέσεις. Θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες για το ποιος μπαίνει σε αυτά τα προγράμματα. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Και ποιον έχουμε από την Επιτροπή? Ε, από την Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ο κύριος Φρανς. Καλησπέρα σε όλους. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμού. Είμαι υπεύθυνο για το Σώμα Αλληλεγγύης και για τη δημιουργία της νέας νομικής βάσης. Θα επανέλθω σε κάποια από τα σημεία τα οποία θίξατε. Πρώτα όμως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια, για τις προτάσεις που κάνατε και τις οποίες σημείωσα. Κατά πρώτον, να επαναλάβω ότι οι ανθρωπιστικές αρχές περιλαμβάνονται στον κανονισμό διασφάλιζοντας τον κανονισμό και να προχωρήσω στο, στην πιο συνήθη ερώτηση για πως αφήνιση που έχει να κάνει με το όριο ηλικία των 30 ετών. Πώς καταλήξαμε σε αυτό το ηλικιακό όριο των 30 ετών. Υπάρχουν τρεις παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, να σας θυμίσω ότι η νομική βάση στη, λειτουργία, στη συνθήκη τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το άρθρο 14.5 που αφορά την συμβολή των νέων Ευρωπαίων στην, Ευρωπαϊκή, στην ανθρωπιστική βοήθεια και τις σχετικές επιχειρήσεις. Είναι η συμβολή δεύτερον, γιατί ακριβώς 30 θα μπορούσε ενδεχομένως να σας ε, ε, προτείνω να διαβάσετε το άρθρο της Επιτροπής για την κατάσταση των νέων ανθρώπων ε, το οποίο εξέδωσε η Επιτροπή το 2018. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο πληθυσμός των νέων Ευρωπαίων φοιτητών έχει σταματήσει ε, ορίζεται στα 29-30 χρόνια που σημαίνει ότι μετά από αυτό το ηλικιακό όριο η μεγαλύτερη, η πλειονότητα των νέων ήδη είναι εργαζόμενοι Επίσης κάτι άλλο που είναι σημαντικό ε, και που φαίνεται στην ενδιάμεση έκθεση του 2017 για το πρόγραμμα εθελοντισμού υπάρχουν ε, σαφείς ενδείξεις ότι υπήρξαν θέσεις ε, στα πρόγραμματα αυτά πάνω από αυτήν την ηλικία. Δεν μπορέσαμε μετά την προκήρυξη των θέσεων αυτών να βρούμε τα κατάλληλα άτομα με τα αντίστοιχα προσόντα. Επίσης, τα δύο τρίτα των εθελοντών που ε, στέλνονται σε αποστολές είναι κάτω από το όριο των 30 και το πιο σημαντικό ε, επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ποιος είναι ο στόχος του πρόγραμματος αυτός. Όπως παρουσιάζουμε τώρα το σώμα ελληνικής δεν εστιάζει σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά υποστήριξη από νέους ανθρώπους στις επιχειρήσεις αυτές. Άρα είναι η εξέλιξη των νέων ανθρώπων. Άρα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα επαγγελματιών και να υποκαταστήσουμε με κάποιο τρόπο τα επαγγέλματα, γιατί ουσιαστικά θα είναι σαν μη πληρωμένη εργασία. Επίσης, να τονίσω και κάτι ακόμα. Ποιους θέλουμε να, ε, σε ποιους θέλουμε να, σε απευθυνόμαστε μάλλον στα προγράμματα αυτά. Έχουμε πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην υπηρεσία θελοντικής, θελοντικής βοήθειας οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι με λίγες δυνατότητες που δεν είναι οι συνείδηστοι οι υποπτοί που συμμετέχουν σε ανταλλαγές, προγράμματα ανταλλαγής μάλλον δεν είναι άτομα που έχουν ε, σπουδές σε καλά πανεπιστήμια αλλά είναι άτομα που ε, δεν έχουν τις δυνατότητες και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Άρα αυτή την πτυχή θέλουμε να λάβουμε υπόψη. Χρειαζόμαστε όμω δύο βασικά βήματα. Μία στρατηγή, την οποία την έχουμε ήδη ε, και που εφαρμόζεται. Χρειαζόμαστε να έχουμε σωστά φορμάτ και επίσης οικονομική στήριξη. Φυσικά το να ε, εμπλέξουμε άτομα από δύσκολες ε, συνθήκες διαβίωσης ε, θα κοστίζει περισσότερο από ότι αν εμπλέξουμε άτομα που θα έχουν εμπειρία από το Πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό είμαστε εμπισμένοι ότι η πρότασή μας, η πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνει υπόψη και δίνει έμφαση στους νέους ανθρώπους ε, Στον υπάρχει μια αναλογία που θα συμπεριλαμβάνει όλους. Και κάτι ακόμα που ρωτήσατε εσείς κυρία Πρόεδρε για τις ε, δραστηριότητες οικοδόμησης ικανοτήτων και για τους τοπικούς οργανισμούς που μπορούν ε, να συμμετάσχουν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση τέτοιου είδους δραστηριότητες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χώρα αλλά έχετε δίκιο εφόσον ε, δίνουμε έμφαση στην νεολαία και αυτές οι δραστηριότητες είναι συμπληρωματικές ε, αυτές οι δραστηριότητες είναι συμπληρωματικές στον αρχικό στόχο ε, του προγράμματος οικονομική στήριξη που δίνουμε στα άτομα. Είπατε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε απλήρωτες ε, μαθητείες ή ε, επαγγέλματα άμυστα. Θα πρέπει να αναλογιστούμε τι σημαίνει θελοντισμός. Είναι κάτι, κάτι που κάνουν οι νέοι χωρίς να πληρώνονται, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά τις βασικές δραστηριότητες που θα πρέπει να επιτελέσει ο οργανισμός και που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του οργανισμού. Είμαστε πολύ προσεκτική στο πώς το πράττουμε αυτό και ενδοευρωπαϊκά, ώστε οι εθελοντές να μην υποκαθιστούν ουσιαστικά επαγγέλματα. Έχουμε λοιπόν εμπειρία σε αυτό εντός της Ευρωπαϊκή Ένωσης και έχουμε και τους συνεδέλφους της ΕΚΟ οι οποίοι αναπτύσσουν παρόμοια προγράμματα ε, με ανθρωπιστική διάσταση. Μιλάμε και για το μέλλον και τη μελλοντική εφαρμογή. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες για τη συμβολή στην ανθρωπιστική βοήθεια και επομένως θα πρέπει να υπάρξουν μορφές πιστοποίησης, προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν την ασφάλεια των ατόμων παρόλο που δεν θα ε, συμμετέχουν σε αποστολέ σε περιοχές όπου υπάρχουν σειράξει. Ελπίζω να απάντησα σε κάποιε από τι ε, ερωτήσει σα και φυσικά αν θέλετε περαιτέρω διευκρινήσει, είμαι πάντα στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την στρατηγική αυτή την οποία εκπονείτε. Δεν λέω ότι θα πρέπει να μείβονται οι νέοι αυτοί, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας χρηματοοικονομικός φραγμός. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό. Ξέρετε ότι α, όλα αυτά τα προγράμματα κοστίζουν ουσιαστικά και υπάρχουν και νέε οικογένειε που δεν έχουν το απαραίτητο οικονομικό υπόβαθρο για να μπορούν να συμμετάσχουν. Είπατε ότι θα πρέπει να προστατεύουμε τους νέους εθελοντές. Δυστυχώς είχαμε και κάποιες περιπτώσεις στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε του δικαιούχου τη βοήθεια αυτή από αυτού που παρέχουν τη βοήθεια αυτή. Δυστυχώ είχαμε και τέτοιε περιπτώσει στο παρελθόν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου των ανθρώπων αυτών, ιδίω αυτών που θα ασχοληθούν για παράδειγμα με τα παιδιά. Υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου, επαλήθευση. Ποιο κάνει την επαλήθευση αυτή, ο ίδιο οργανισμό, ο οποίο απασχολεί αυτού του θελοντέ. Κοιτάξτε, μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύης έχουμε και μια καινοτομία. Στο παρελθόν βασιζόμασταν πάρα πολύ στους επιτόπου οργανισμούς, οι οποίοι ήταν επιστοποιημένοι βέβαια ή είχαν ένα απαραίτητο σήμα ποιότητος, οι οποίοι οι ίδιοι έλεγχαν ότι οι εθελοντές που απασχολούσαν είχαν ε, όχι μόνο τα απαραίτητα κινήτρα, αλλά ότι είχαν και τις δεξιότητες και τα προσόντα προκειμένου να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες καταστάσεις και προκειμένου να εργαστούν με συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Το σύστημα τώρα έχει αλλάξει και παρέχουμε εμεί μια μεγαλύτερη υποστήριξη. Αυτοί οι νέοι εθελοντέ πρέπει εκ των προτέρων να καταχωρήσουν στο, στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη τα στοιχεία του, τι δεξιότητέ του και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να περάσουν και από ένα σύστημα επιγραμμική κατάρτιση προτού φτάσουν στο σύστημα τη απευθεία κατάρτιση προβλέπετε. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε λίγο να βλέπουμε ποιον δρόμο μαθητείας, σπουδών και τα λοιπά έχουν ακολουθήσει οι νέοι αυτοί προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες. Βέβαια, ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως το να εργάζεται κανείς ε, με παιδιά ή ε, αυτό προβλέπεται πολλές φορές ε, ακόμα και στην παροχή βοήθειας προς τα παιδιά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου πάλι προβλέπεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επαλήθευσης του προφίλ και των ικανοτήτων. στην ε, δική μου την πόλη προκειμένου να μπορώ για παράδειγμα να εργάζομαι στο σχολείο της πόλης μου θα πρέπει να περνάω από ένα σύστημα επαλήθευσης ακόμα και του ποινικού μου μητρώου. Το σημαντικό είναι να μην προστατεύουμε μόνο τους εθελοντές που στέλνουμε, αλλά και τους δικαιούχους της ανθρωπιστικής αυτής βοήθειας. Απευθύνομαι τώρα στην Ελένη, δεν ξέρω αν θέλεις ε, να προβεί σε κάποιες παρατηρήσεις, κάποια συμπεράσματα, πρωτού κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έκτος μικροφώνου. Πριν ευχαριστήσω τον Κρίστιαν που βοήθησε πολύ στη σύνταξη του κειμένου, στην... το παρέλειψα προηγουμένως, το ξέχασα μάλλον, Α, θα ήθελα να σας πω και τα εξή. Συμφωνώ με αρκετά από αυτά που έχουμε ακούσει από την Επιτροπή και από τους συναδέλφους, τον συνάδελφο Γκερέρο, ε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα πνεύμα και μια κουλτούρα εθελοντισμού. Αυτό είναι ένας βασικός στόχος της όλης προσπάθειας. Αλλά δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα στρατό μισθοφόρων εθελοντών. αυτοί που θα εργάζονται στην εθελοντική διαδικασία θα πρέπει να έχουν και την δουλειά τους και την σταδιοδρομία τους και όταν χρειαστεί να πάνε σε ένα πεδίο να μπορούν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους και να πάνε να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Α, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να λειτουργήσουν μέσα σε όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα. Άρα εφόσον θα αφήσει τη δουλειά του θα πρέπει και να πληρώνεται όταν θα φτάσει. Τουλάχιστον να του καλύπτονται κάποια έξοδα. Ε, γι' αυτό είπαμε ότι απαιτούνται κάποια κονδύλια για την λειτουργία του σώματος. Ε, επίσης, τα κονδύλια δεν θα πρέπει να διατίθενται για ένα υδροκέφαλο ε, διοικητικό σώμα με ελάχιστα κονδύλια για το πεδίο. Απέναντίας θα πρέπει να είναι τα πολλά ποσά να πηγαίνουν στο πεδίο και τα λίγα να παραμένουν στην διοίκηση. Θέλω να σας πω ότι έχει πολύ δίκιο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που λέει ότι όσο πιο πολλές σπουδέ έχει κάποιος τόσο πιο λίγες πιθανότητες έχει να ε, εμπλακεί στον ε, εθελοντισμό αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω από την προσωπική μου εμπειρία που έχω λάβει μέρος σε τουλάχιστον 150 ε, αποστολές ότι στις εμπόλεμες ζώνες δεν υπήρξε εθελοντής που να ήρθε δύο φορές. Δηλαδή για μία φορά θα έρθει ένας εθελοντής, αλλά δεύτερη φορά δεν έρχεται, ειδικά στις εμπόλεμε ζώνε. Άρα το να δημιουργήσουμε ένα στρατό 100.000 εθελοντών δεν νομίζω ότι θα είναι και ε, ε, μια δυνατότητα μέχρι το 2020. Όπως και να έχει το θέμα, σας ευχαριστώ πολύ και θα ειδούμε παραπέρα τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου, 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Ας περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της μίλησης διάταξης, ώρα των ερωτήσεων. Δύο ερωτήσεις έχουμε εδώ πέρα για την Επιτροπή μας. Η πρώτη είναι μία ερώτηση από την υποφαινόμενη Απευθύνουμε εδώ πέρα στον επικεφαλής των σχέσεων με το Αφγανιστάν και εμπλέκεται εδώ πέρα η κυρία Σαρτζεντίνη όσον αφορά τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν. Πριν από την διάσκεψη του 2016 για το Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο που έφερε τον τίτλο «Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν». Στο παράρτημα λεγόταν ότι θα υπήρχε μια δέσμη επανένταξης προκειμένου να μπορούν οι υπήκοοι του Αφγανιστάν που βρίσκονται σε τρίτες χώρε να επιστρέψουν στη χώρα του στο Αφγανιστάν. Εμεί θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι έγινε τελικά με το πρόγραμμα αυτό, ποια ήταν η χρηματοδότηση, που πήγανε τα χρήματα που επικεντρώνεται το πρόγραμμα αυτό, έχει να κάνει κυρίως με Αυγανού οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και επιστρέφουν στο Αφγανιστάν ή έχει να κάνει γενικότερα με την επανένταξη προσφύγων από όμορε χώρε όπως το Ιράν και το Πακιστάν. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένω είναι εδώ για να απαντήσει. Ζων Λουιβίλ, παρακαλώ. Σα είδα να μπαίνετε και δεν ήξερα για ποια ερώτηση ήταν αρμόδιος. Ο Ζων Βίλ, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όντω, μπορεί να σας προκανεί έκπληξη ξαφνικά ότι είμαι αρμόδιο για την Ασία, όχι για το Αφγανιστάν, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Λοιπόν, να υπενθυμίσω πολύ γρήγορα το θέμα το οποίο ετέθη. Δεν θα μπω σε λεπτό μέρη. σε καμία περίπτωση. Θα ήθελα να σας δώσω πολύ γρήγορα μία απάντηση. Θα μπορούσα τέλο πάντων να μακρηγορήσω αρκετά. Ενδεχομένω γραπτό θα μπορούσατε να μα δώσετε την πιο λεπτομερή απάντηση. Νομίζω το καλύτερο θα ήταν γραπτό να μα δώσετε την απάντησή σα από ότι θα μα διαβάσετε τώρα του αριθμού. Σε κάθε περίπτωση θα υποβάλω και το γραπτό κείμενο το οποίο περιέχει πολλά αριθμητικά δεδομένα τα οποία είναι σημαντικό να έχετε για να καταλάβετε ποιου υπολογισμού έχουν γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε συνολικά στο πρόγραμμα αυτό επανένταξη των Αυγανών 194 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το συνολικό ποσό το οποίο δόθηκε, χρηματοδοτείται από το DCI πλήρως. Από το μέσο δηλαδή αναπτυξιακής βοήθειας. 131 εκατομμύρια τώρα από αυτά και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα ευρώ έχουν ε, προγραμματιστεί μέχρι σήμερα. Τώρα το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί το πρώτο ήμιση του 2019. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα όσον αφορά την εφαρμογή. Το συνολικό ποσό το οποίο έχει εκταμιευτεί είναι 57 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το μερίδιο των κονδυλίων ανάμεσα στα τρία αυτά σκέλη τα οποία προβλέπονταν στο πρόγραμμα Joint Way Forward για το Αφγανιστάν είναι ως εξή. Πρώτον, δέσμη κινήτρων 39 εκατομμύρια ευρώ επανένταξη μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και σχετικά σχέδια 18 εκατομμύρια ευρώ και το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της απασχόλησης 21 εκατομμύρια ευρώ. Πέρα από τα τρία αυτά στοιχεία τα οποία εντοπίζονται ξεκάθαρα στο πρόγραμμα αυτό Joint Way Forward, έχουμε εκταμιεύσει περίπου 53 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και προστασία, καθώς επίσης και στην κατανομή γεών για τους επιστρέφοντες στο Αφγανιστάν και τις κοινότητές τους. Όλες αυτές οι δράσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζονται σε πραγματικέ ανάγκε και έχουν ω στόχο την επανένταξη και την επιστροφή όλων των Αφγανών υπηκών ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκονταν. Όσον αφορά τώρα του Αφγανού υπηκόου που βρίσκονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνεται υπόψη και η χρηματοδότηση που έχει δοθεί από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Μολονότι υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγε από το Ιράν και το Πακιστάν, ιδίω τα τελευταία χρόνια, και καθότι εντοπίζονται εκεί πέρα υψηλότερε ανάγκε, οι δικαιούχοι του προγράμματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για του ανθρώπου λοιπόν που έρχονται από το Ιράν και το Πακιστάν, αλλά και για του εσωτερικά εκτοπισμένου στο Αφγανιστάν, περίπου 96%, 96 των δικαιούχων είναι αυτοί. Και βέβαια έχουμε και τους ε, Αφγανού υπηκόους που έρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστοιχούν περίπου στο 4%. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων από τον Οκτώβριο του 2016, τότε δηλαδή που υπεγράφει το πρόγραμμα Joint Way Forward, είναι πάνω από 21.000 υπήκοοι. Αναφέρομαι σε αυτούς που επιστρέφουν βέβαια πάντα στο Αφγανιστάν. Προβλέπεται επίση λοιπόν ότι θα υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση για να έχουν οι άνθρωποι αφήτα προ το ζήν, τι απαραίτητε ευκαιρίε ένταξη στην αγορά εργασία, πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτιση και εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και δημιουργία ικανοτήτων για όλε τι αρμόδιε αρχέ, προκειμένου να εφαρμόσουν το απαραίτητο πλαίσιο πολιτική για την υλοποίηση του προγράμματος. Περίπου 500.000 είναι οι άνθρωποι αυτοί, περίπου μισό εκατομμύριο λοιπόν, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιστροφή και την Επανένταξη. Υπάρχουν πολλοί εταίροι οι οποίοι εφαρμόζουν το πρόγραμμα αυτό, Παγκόσμια Τράπεζα, η UNICEF, το πρόγραμμα για το ενδιέτημα των Ηνωμένων Εθνών, η ITC, η DRC, και υπάρχουν και πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει, τι οποίε δεν θα παριθμίσω αυτή τη στιγμή. Η υποστήριξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνεται κυρίω στον τομέα τη σταθερότητα και τη ασφάλεια. Οι δραστηριότητε για την επανένταξη έχουν οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Ε, η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρησιμοποιείται προκειμένου να μετριαστούν πιθανοί κίνδυνοι όσον αφορά την ε, σταθερότητα. Σας έδωσα, αν θέλετε, σε πολύ γραμμέ ε, την βασική απάντηση στο ερώτημό σα αυτό. Δεν θα ήθελα να σα χωρίσω αυτή τη στιγμή με ιδιαίτερα λεπτομερή αριθμητικά δεδομένα, γιατί θα περιπλακούν πάρα πολύ τα πράγματα και προφανώ θα σα ε, υποβάλλω το κείμενο αυτό, καθώ επίση και περισσότερε λεπτομέρειε γραπτό, κυρία Πρόεδρε, προκειμένου να μπορέσετε να τα μελετήσετε αυτά επαρκώς. Πρόεδρο, Σα ευχαριστούμε πολύ. Μία ερώτηση έχω για τα αριθμητικά δεδομένα τα οποία μα δώσατε ενδεχομένω να καλύτερα να διαβάσω και το κείμενό σα. Είπατε 21.000 έχουν ήδη βοηθηθεί. Ισχύει αυτό. Να αναφέρομαι σε ανθρώπου που επέστρεψαν στο Αφγανιστάν. Το 4% αυτών, μόνο 4% προέρχεται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το 96% των επιστρεφόντων είναι από τις όμορε χώρες, από το Ιράν, το Πακιστάν, καλά κατάλαβα. Και είπατε 500.000, ποιοι είναι αυτοί. Να προσθέσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. 21.000 Ιράν, Αφγανιστάν και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στο Αφγανιστάν, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας. Οι 500.000 είναι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που εποφελούνται από τη γενικότερη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο από το πρόγραμμα της επανένταξης, αλλά και από όλα αυτά τα προγράμματα υποστήριξης για τις Διάφορε κοινότητε στο Αφγανιστάν για την δημιουργία δυνατοτήτων, για την τεχνική υποστήριξη. Αν λάβουμε υπόψη του δικαιούχου για όλα αυτά τα προγράμματα, φτάνουμε του 500.000. Πολύ ωραία, λέει πρόεδρο. Εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα να πάρει το λόγο. Η Σοντάλ Μαρινή δεν είναι παρούσα, είναι εδώ. Όχι, δεν τη βλέπω. Για το επόμενο, για το επόμενο ερώτημα είναι αρμόδια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πλήρης η απάντηση από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και θα θέλαμε και ένα αντίγραφο της απάντησής σας ή δυνατόν. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τα δάση. Um, ρωτάει η κυρία Χάουταλα για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου, στο οποίο ζητάμε από την Επιτροπή για ένα σχέδιο δράσης για τα δάση. Ήταν καλή εισαγωγή σας. Λοιπόν, στην έκθεση που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο, που ανέκρινε το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο, για τη χρήση των πόρων συγκεκριμένα για τα δάση, το Κοινοβούλιο ρώτησε την Επιτροπή να ε, προβεί σε μία μελέτη αντικτύπου και να ε, κάνει διαβούλευση με τη διαφερόμενα μέρη, με άτομα από τις τοπικές κοινότητες για να δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στην ε, αποδάση και την υποβάθμιση των δασών που θα περιλαμβάνει και ένα μηχανισμό παρακολούθησης για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν ε, χρηματοδοτικέ ε, συναλλαγέ ε, που σχετίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την αποψήλωση και την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης να προαχθούν να προαχθεί τεχνική στήριξη στις τοπικές κοινότητες. Πώς έχει σκοπό λοιπόν η Επιτροπή να προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Ποιος θα απαντήσει Δεν έχω το όνομά σας, αλλά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σαν Ταλμαρή, έχετε δίκιο. Αλλά είμαι στην μονάδα της και συγκεκριμένα στον τομέα των δασών. Πρώτα απ' όλα η Επιτροπή είναι ευχαριστημένη με το ψήφισμα του Κοινοβουλία για τη διαφανή ε, διαχείριση των δασών. Όσον αφορά το θέμα της αποψήλωσης, η Επιτροπή, όπως και το Ευρωκοινοβούλιο, θεωρεί ότι είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που χρειάζεται μια ε, ολοκληρωμένη και διατομεακή ανταπόκριση η αποδόμηση των δασών αποτελεί ένα βασικό στοιχείο των εργασιών της Ευρωπαϊκής στην εφαρμογή της Ατζέντα 2030 ε, για την βιώσιμη ανάπτυξη και στο πλαίσιο φυσικά της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά την Ατζέντα 2030, και την αξιολόγηση που έχει γίνει για την αποδάσωση στις τρίτες χώρες και η άλλη μελέτη που έγινε για τη δημιουργία σχεδίου δράσης της Βρυξέλλωσης για την αποψήλωση που εκδόθηκε το 2018. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν η Επιτροπή προτίθεται να εντεθειοποιήσει τις εργασίες για να καταπολεμήσει την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών. Αυτή η ανακοίνωση της Επιτροπής θα έχει ως στόχο να ε, ανακοινώσει, να γνωστοποιήσει μάλλον τη δράση που έχει αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ε, να δείξει ποια είναι τα σχετικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμή και επίση ε, να γίνουν και διαβουλεύσεις μελλοντικά με την κοινωνία των πολιτών, τα κράτη-μέλη ε, για, το, για τις δράσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο πολιτικών για την αποδάσωση. Το 2017 η Γενική Διεύθυνση ε, Περιβάλλοντος ε, διεξήγαγε μία, ε, μία εκδήλωση για την παράνομη και το εμπόριο. Επίσης θα γίνουν διαβουλεύσεις για να έχουμε τις απόψεις του κοινού. Αυτά. Okay. to... Μάλιστα, Χάιντι, κάτι άλλο θες να ρωτήσεις. Ναι, ναι, λίγο εν συνεχεία των όσων υπόθηκαν. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα ότι η διαβούλευση αυτή θα ξεκινήσει σύντομα και ελπίζω ότι θα οδηγηθούμε σε κάποια αποτελέσματα από τη διαδικασία αυτή ήδη στα πλαίσια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Τι σχεδιάζετε λοιπόν εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπετε κάτι πριν το τέλος της θητείας αυτής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Αυτό ελπίζουμε. Για να αποσαφηνίσω λίγο και τα πράγματα. Περιμένουμε ακόμα, θέλετε, την έγκριση, το πράσινο φως από την ε, Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ξεκινήσουμε τη σχετική εργασία. Ήδη έχουμε αρχίσει βέβαια να επεξεργαζόμαστε το όλο ζήτημα, παρόλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, συγκεκριμένε διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Πρέπει εμείς καταρχάς να εκπονήσουμε τον οδικό χάρτη για την ανακοίνωση αυτή. Αυτό θα μας πάρει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή όμως ο οδικός χάρτης ανακοινωθεί, αφού περάσουν δηλαδή τέσσερι αυτέ αυτές εβδομάδες, τότε μόνο μπορεί να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος μας είναι η ανακοίνωση αυτή να είναι έτοιμη πριν το 2019, αλλά αυτό και πάλι θα εγκριθεί από το πότε θα πάρουμε αυτό το πράσινο φως στην αρχική έγκριση που σας είπα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να στο ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό. Χάιντι, συμφωνείτε? με την άδειά σα, κυρία Πρόεδρε, ένα σύντομο επιμέρου ερώτημα. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν και διάφορα κράτη-μέλη που μέσω τη δήλωση εταιρική σχέση του Άμστερνταμ έχουν ζητήσει το ίδιο πράγμα. Το ίδιο έχουν κάνει και πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με το ζήτημα της υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως άλλωστε αναφέρεται και στη μελέτη σκοπιμότητος την οποία αναφέρεται πολύ γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος, με ένα ναι ή όχι δυνατόν, γιατί πρέπει πραγματικά να ολοκληρώσουμε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως σας είπα, βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο και δεν μπορώ να γνωρίζω ακόμα αυτή τη στιγμή τι θα συμπεριληφθεί στη μελλοντική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση πάντως βασιζόμαστε στα πορίσματα της μελέτης κοπιμότητος. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προς την Χάιντι και τους άλλους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της δασικής νομοθεσίας, Αύριο το βράδυ προβλέπεται μία εκδήλωση για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που υπερασπίζονται επίσης και τα δάση και τη σχετική νομοθεσία. Θα έχουμε λοιπόν και ανθρώπους από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ που θα μας μιλήσουν για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδίω στον περιβαλλοντικό τομέα. Και αύριο το πρωί όμως υπάρχει μια αντίστοιχη εκδήλωση, λέει η κυρία Χάιντι Χάουταλα. Όπως θα θυμάστε, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση όσον αφορά την βιωσιμότητα και τη διαφάνεια Τη εφοδιαστική αλυσίδα για τον καφέ και το κακάο. Τον Ιούλιο έγινε αυτό. Αύριο το πρωί θα φιλοξενήσουμε μια εκδήλωση στις 9.30 το πρωί όσον αφορά την, τις νομικές δεσμευτικές υποχρεώσεις που υπάρχουν όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα για το κακάο και ιδίως τη συμμετοχή των παιδιών ως εργαζόμενοι σε αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έρθει και στην εκδήλωση αυτή γιατί οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θέλουν και στον τομέα αυτό να υπάρχει πλέον ένα δεσμευτικό εργαλείο, ένα δεσμευτικός μηχανισμός. Αύριο λοιπόν έχουμε και μία εκδήλωση από τις 3 ως τις 5 στην SP3 ή 3 και αύριο έχουμε μια εκδήλωση με την Επιτροπή Άγκρη, κοινή συνεδρίαση για να ακούσουμε τις, τα πορίσματα της παγκόσμιας διάσκεψης όσον αφορά τον υποσυτισμό από τις 5.30 έως τις 6.30 αύριο προβλέπετε αυτό. Ενδεχομένως να σας στείλουμε και ένα email για να σας ενημερώσουμε για τις εκδηλώσεις αυτές. Δεν έχουμε τίποτα από τα διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση, καλύτερα να μην σας δώσουμε ημερομηνία γιατί παντού λέγεται ενδεχομένως. Ε, 10 Δεκεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου ενδεχομένω. Θα δούμε. Α, έχει επιβεβαιωθεί. Έχουμε και το βραβείο Ζαχάροφ, μάλιστα. Άρα σίγουρα στις 10 Δεκεμβρίου για την παρουσίαση τη σχετική με το βραβείο Ζαχάροφ, από κοινού βέβαια με την Επιτροπή ΑΦΕΤ, εξωτερικών υποθέσεων. Ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό η συνεδρίαση. Σε λίγο θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Νομίζω ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Λοιπόν, διακόπτουμε για πέντε περίπου λεπτά και θα συνεχίσουμε μετά με τους συντονιστές. Σας ευχαριστώ.